προσβλέπουμε στο προτάσεις πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μελλοντικό μηχανισμό ε, επίλυσης της κρίσης τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Now Κύριε Κέλλαμ, πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και θα δώσω το πρώτο το λόγο στην κυρία Μπασέσκου.